Καλημέρα, ξεκινάει η Σύνοδος. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι μια προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τον κανόνα ε, της ε, μοναδικής χειραποσκευής που επιβάλλουν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες. Ο κύριος Σίμψον, που είναι ο συγγραφέας, έχει πέντε λεφτά για να μας παρουσιάσει την ερώτηση. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε ήδη, γιατί δεν είναι εδώ εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Αξίζει τον κόπο. I Ούτως ή άλλως, όλη η ουσία είναι προς την προφορική ερώτηση που θέλουμε να απευθύνουμε στην Επιτροπή. Αν δεν είναι Επιτροπή, δεν τι νόημα έχει. Ο Επίτροπος έρχεται. Εγώ εκπροσωπώ την ε, Επιτροπή Μεταφορών. Ίσα παρουσιάζω αυτή την ε, προφορική ερώτηση, η οποία αφορά την ε, υποχρέωση μίας και μόνο χειραποσκευής που επιβάλλουν σε αεροπορικές εταιρείε. Η Επιτροπή μου θεωρεί ότι πρέπει να αναλάβουμε θράση για να αντιμετωπίσουμε την ασυνέπεια και την έλλειψη διαφάνειας που συχνά αντιμετωπίζουν οι επιβάτες όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Είναι κλασική πρακτική εδώ και χρόνια, Πρόεδρε, ότι οι επιβάτες μπορούν να αγοράζουν ε, κάποια πράγματα ε, στο αεροδρόμιο και αυτά να τα παίρνουν δωρεάν ε, στις χειραποσκευές τους. η εισαγωγή τελών για αυτές τις αγορές τώρα, καθώς και τέλη για έξτρα χειραποσκευές όπως οι τσάντες που περιέχουν τους προσωπικούς υπολογιτές, αυτό είναι το θέμα. Σε ορισμένε αεροπορικέ εταιρείε, ακόμα και ένα μπουκάλι ουίσκι ε, του επιβάλλεται τέλο. Ενώ σε άλλε αεροπορικέ εταιρείε αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει μια συνέπεια λοιπόν. Υπάρχει έλλειψη διαφάνεια στο τι συμβαίνει στι αεροπορικέ εταιρείε. Και αυτή η έλλειψη συνέπεια μα ανησυχεί. Πιστεύουμε ότι κάποιες ευρωπαϊκές ε, εταιρείες αδιαφορούν για τις κατευθυντήριες γραμμές της ε, οργάνωσης πολιτικής αεροπορίας που έχει αρνητικές επιπτώσεις και στους επιβάτες και στο λιανεμπόριο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι κανόνες για τις χειραποσκευές θα πρέπει να ακολουθούν κάποιους, ε, να έχουν κάποια συνέπεια. Και καταλαβαίνω βεβαίως και τα εμπορικά ωφέλη για τις Αεροπορικέ εταιρείε. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια κάποιες αεροπορικές εταιρείε θέλησαν να επιβάλλουν κάποιο τέλος, να κάνουν του επιβάτες να πληρώνουν για τα πάντα, ενώ κάποιες άλλες όχι. Και ο τρόπος που επιβάλλουν το οποιοδήποτε τέλος, που χρεώνουν οτιδήποτε, ε, είναι προβληματικός, γιατί θέλω το κοινό να αντιμετωπίζει μια κατάσταση διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για την ευρωπαϊκή αεροπορία και συχνά ε, προκαλεί θυμό και σύγχυση στους επιβάτες. Και οι επιβάτες έχουν την αίσθηση ότι τους κλέβουν οι αεροπορικές εταιρείες. Αυτό είναι πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Ντεχούχτ. Uh, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, Καλημέρα σας. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και επισημάνει και στην ερώτησή του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι οι συνθήκες ε, που, αφορούν τις χειραποσκευές ε, και ο βαθμός αυστηρότητας ε, ποικίλει από αερογραμμή σε αερογραμμή. Παρόλο που υπάρχουν νέες διατάξεις, δεν εφαρμόζονται παρόμοια. Βέβαια είναι πολλές υπηρεσίες ε, που προσφέρονται στους ε, επιβάτες σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Η ελευθερία των ε, αεροπορικών εταιριών να κανονίσουν τα τέλη των αεροπορικών εισιτηρίων και γενικώ τα τέλη είναι ένας από τους λόγους της, της συνθήκης της ενιαίας αγοράς των ενιών εθέρων. Και έτσι μειώθηκαν οι τιμές λόγω του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και επιβατών. Οι αεροπορικές εταιρείες ελεύθερα μπορούν να προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους βέβαια με διαφανή τρόπο και ε, τηρώντας την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις αεροπορικές υπηρεσίες. Ε, γιατί έχουμε τον κανονισμό 82 του 2002 ε, για την ευθύνη των αεροπορικών εταιριών σε περίπτωση αεροπορικών ατυχημάτων. Και έχουμε και ένα κανονισμό του 2008 εφόσον λειτουργήσει η εύρυθμα η αγορά και υπάρχει διαφανής ενημέρωση, μπορεί αυτό να γίνει κριτήριο για την επιλογή της ΑΒ αεροπορικής εταιρείας. Ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Οι επιβάτες δικαιούνται να γνωρίζουν εκ των προτέρων και με διαφάνεια τις ε, αρχές που ισχύουν για τις χειραποσκευές. Οπότε με την καλύτερη ενημέρωση στους επιβάτες, το θέμα της ανομιμορφίας των διατάξεων ε, για τις χειραποσκευές μπορεί να καλυφθεί. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Ο ρόλος των ε, εθνικών αρχών ε, επιβολής της νομοθεσίας θα πρέπει να θεωρηθεί ως τμήμα της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών που η αναθεώρησή της θα παρουσιαστεί στο πρώτο εξάμεινο του 2013. Η πολιτική της μίας και μόνο χειραποσκευής επηρεάζει και τα συμφέροντα των ε, ε, καταστημάτων ε, αφορολογήτων στα αεροπόρια. Θα πρέπει να ενημερώνονται φυσικά οι πολίτες και οι διατάξεις αυτές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν τους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν στα αεροδρόμια. Ευχαριστώ. Μιλούν οι εκπρόσωποι των ομάδων. Ο κύριος Μπάχ από το ΕΛΚ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ από τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Ελκαντράουι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ από τους ε, φιλελεύθερους. Ο κύριος Έντουαρτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. What items are essential and non-essential, the counting. Θα, θα πρέπει ε, να δούμε τι ισχύει στις, περι... στις περιπτώσεις αυτές. Δυστυχώς υπάρχουν ε, διατάξεις που εφαρμόζονται πολύ διαφορετικά από κάθε αεροπορική εταιρεία ή από κάθε αεροδρόμιο σε ό,τι αφορά τις χειραποσκευές αλλά και τις αγορές ε, στο... στα καταστήματα ελληνικής στο αεροδρόμιο. Δεν υπάρχουν ενίοι κανόνες, υπάρχει μια σύγχυση που δημιουργεί προβλήματα και ενοχλεί τους επιβάτες. Έχουμε τελικά σε μείωση των πωλήσεων λιανική στα αεροδρόμια εξαιτία αυτή τη σύγχυση και τη έλλειψη ενημέρωση. Είναι υπερβολικέ ε, και αυθαίρετε πολλέ φορέ ε, ε, οι διατάξει και οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι αεροπορικέ εταιρείε Για να μην πω ότι είναι και κομικοί μερικέ φορέ αυτοί οι περιορισμοί. Επίση είναι ένα άμεσο τρόπο τιμωρία και επιβολής προστήμων στους επιβάτε από το προσωπικό εδάφος. Μερικέ φορέ καταπατώνται και οι διατάξεις ε, του δικαίου ανταγωνισμού. Πιστεύω θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κοινή λογική για το ποιο είναι το κατάλληλο μέγεθο ε, και το βάρο τη χειραποσκευή. Και καλό θα ήταν να τεθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινά ανώτατα όρια για του περιορισμού. Νομίζω ότι έτσι θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη σαφήνεια για τι αποσκευέ αλλά και για τι αγορέ στα καταστήματα λιανική. Θα πρέπει να προστατεύσουμε του επιβάτε και να του επιτρέψουμε να έχουν λογικές χειραποσκευές ε, και να μπορούν να αγοράζουν κάποια προϊόντα από τα καταστήματα ελληνικής. Χρειαζόμαστε κάποια ενιαία μέτρα. Δεν θα πρέπει ε, να είναι μόνο διατάξεις της θεωρίας, να εφαρμόζονται και πράγματος και να μην αφήνουμε τους επιβάτες ε, στο έλεος των αεροπορικών εταιριών ή στο προσωπικό εδάφους στις πύλες εξόδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τους πράσινους, κυρία Λίχτεμπέργκερ, για 1,5 λεπτό.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 το ECR ο κύριος Βλάσακ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι διακοπές μπορεί να γίνουν ε, περίπλοκες και δαπανηρές λόγω των χειραποσκευών και των αποσκευών γενικά. Μπορεί να γίνει μια δυσάρεστη εμπειρία. Ε, μερικές φορές έχουμε καθυστερήσεις λόγω των αποσκευών που δεν φτάνουν ή δεν φτάνουν καν ποτέ. Τώρα για τις χειραποσκευές, ε, κάποιες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν δωρεάν ε, μεταφορά χειραποσκευών μέχρι κάποιο μέγεθος. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως επιβάλλουν στους επιβάτες να τις δώσουν στο check-in και μερικές φορές επιβάλλουν τέλη. Θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις ε, στις αεροπορικές εταιρείες να επιβάλλουμε κάποιους εναρμονισμένους κανόνες. Οι επιβάτες πρέπει να έχουν ελευθερία επιλογής κυρίως μερικές ε, μεταξύ διαφόρων μεταφορικών εταιριών. Οι εταιρείε low cost είναι φθηνέ, αλλά δίνουν και λιγότερες υπηρεσίες. Νομίζω ότι μερικές φορές ε, Έχουμε προβλήματα. Ξέρουμε ότι κάθε νέο κανονισμός βέβαια ε, δημιουργεί επιπλέον κόστος για, τους, ε, ε, για τις εταιρείε. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε υπερβολικό επιπλέον κόστος για τις εταιρείε. Ο κύριος Μέρφυ από την ΚΟΕ για ένα λεπτό. Υπάρχει μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην επιβάνητη και την, εταιρική, και την αεροπορική εταιρεία. αλλά δεν είναι σχέση ίσων πολλοί ε, επιβάτες δεν έχουν καμία επιλογή παραπάνω παρά να πάρουν μια συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Και πολλέ ε, εταιρείε χρησιμοποιούν αυτόν τον κανόνα όχι προ το συμφέρον των επιβατών, αλλά σαν μέσον για να αυξήσουν τους, τα κέρδη τους επιβάλλοντας ε, διογκωμένα τέλη στους επιβάτες για να δώσουν στο check-in τις αποσκευές τους. Ξέρουμε ότι αυτό είναι μία από τις πολλές άγριες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εταιρείε για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Και βεβαίως ε, ποιος είναι εδώ στο, στον προμαχώνα, η Ryanair, ε, που κλέβουν τους ε, επιβάτες, επιβάλλουν επιπλέον τέλη στις πιστοτικές κάρτες κτλ. Πρόκειται για καπιταλιστική απληστία που σκοπό έχει να μεγιστοποιήσει το κέρδος πάση θυσία. Η αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν με δικτατορικό τρόπο. Μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Θα κάνετε τίποτα ή εν πάση ξέρετε αν η Ιρλανδική κυβέρνηση θα κάνει τίποτα και θα τιμήσει την υπόσχεσή της ε, για να κάνει κάτι για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταντάν για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η πολιτική της ε, χειραποσκευής δεν είναι μια απλή εμπορική πολιτική όπως οι υπόλοιπε. Θα, τους, ε, θα υποχρεώσει τους επιβάτες να κάνουν α, συγκεκριμένες επιλογές. Δηλαδή, αντί να αγοράσουν στα καταστήματα ελληνική αεροδρόμια, υποχρεούνται να αγοράσουν μέσα στο αεροπλάνο. Δεν είναι σαφής η πολιτική κύριε Επίτροπε και τα μέτρα περιορισμού για τις χειραποσκευές και τις αποσκευές εφόσον είναι δραστικά ε, καταστρατηγούν την ελευθερία των επιβατών δεν έχουν δικαίωμα επιλογή, δεν έχουν δικαίωμα αγορά προϊόντων στα καταστήματα ελληνική αεροδρόμια, αλλά έχει κάτι τέτοιο επιπτώσει και στα αεροδρόμια και ιδιαίτερα στα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Στα αεροδρόμια αυτά, τα περιφερειακά, τα προβλήματα είναι πολύ ανησυχητικά. Οι εταιρείε low cost ε, εγκαθίστανται σε αυτά τα μικρά αεροδρόμια και οι ίδιε εταιρείε εφαρμόζουν πολιτικέ αποσκευών που ε, βλάπτει τα συμφέροντα των αεροδρομίων. Ε, υπάρχει κίνδυνος λοιπόν εξάρτηση των περιφερειακών αεροδρομίων από τις εταιρείε low cost. Θα πρέπει να καταδικάσουμε τα αεροδρόμια αυτά να δεχτούν ανεφόρον όλες τις ε, προϋποθέσεις και τους όρους των αεροπορικών εταιρείων και εις βάρος των επιβατών. Αυτό το διαπιστώσαμε με την επέλαση των εταιριών low cost στα περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν θα πρέπει να έχουμε κατάχρηση δεσπόζων θέσει από τι αεροπορικέ εταιρείε και η πολιτική τη μη χειραποσκευή δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ των αεροπορικών εταιριών. Υπάρχει κίνδυνο να καταστρατηγηθεί ο θεμητό ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι χρειάζεται τουλάχιστον τα φορολόγια τα προϊόντα να μην θεωρούνται χειραποσκευέ. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε μόνο να αντιμετωπίσουμε δραστικά το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγέλα Σέντερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να επισημάνω την κακώς εννοούμενη εμπορική ελευθερία και την αναγκαία ε, τήρηση των δικαιωμάτων των επιβατών που βρίσκονται σε σύγχυση μεταξύ της αδιαφάνειας των τιμών, έλλειψης ενημέρωσης και τεράστιες δυσκολίες για διαμαρτυρία και ένσταση. Έχουμε πολλές καταχρήσεις για να μην πω και κακή μεταχείριση από το προσωπικό εδάφος των αεροπορικών εταιριών που υπό την πίεση των αεροπορικών αυτών εταιριών ε, κακομεταχειρίζονται τους επιβάτες, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους. Οι γυναίκες χρειαζόμαστε μία επιπλέον τσάντα. Εκεί έχουμε τα έγγραφά μας, ε, τα διαβατηριά μας. Θεωρείται μία επιπλέον χειραποσκευή. Και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα έχουμε στα περιφερειακά αεροδρόμια που υφίστανται τον εκβιασμό των αεροπορικών εταιριών. Μόνο με περισσότερη ενημέρωση, όπω είπατε κύριε Επίτροπε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αλλά δεν αρκεί ούτε αυτό, γιατί έχουμε αντιφατικέ ε, διατάξει. Χρειαζόμαστε ομοιογενεί, ομοιόμορφου και σαφεί κανόνε. Η Ισπανική νομοθεσία διευκολύνει και προστατεύει τον επιβάτη, αλλά εκεί επικαλούνται οι εταιρείε ε, το επιχείρημα της ασφάλειας και του μονοπωλίου που έχουν στα περιφερειακά αεροδρόμια για να συνεχίσουν αυτή την πολιτική κατάχρηση. Θέλουμε μία εναρμόνιση, ομοιόμορφους κανόνες. Μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε την ισότητα των επιβατών και θα μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Κύριος Κράμερ, για ένα λεπτό. κύριος Φιντάντσα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι κανόνες για τη μεταφορά χειραποσκευής, όπως εφαρμοζόταν μέχρι στιγμής, οδηγούν σε διαφορετικές καταστάσεις. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείε επιβάλλουν υπερβολικούς περιορισμούς αδικαιολόγητους και περιορίζουν τη δυνατότητα αγοράς αγαθών από τους επιβάτες, ειδικά στο εσωτερικό του αεροδρομίου. Επομένως περιορίζονται έτσι τα δικαιώματα των επιβατών και ε, προωθούν τις επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Ε, καμιά φορά έχουμε σημαντικές απώλειες όμως για το λιανεμπόριο του αεροδρομίου. Ε, και κυρίως έχουμε πρόβλημα στα περιφερειακά και μικρότερα αεροδρόμια. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει διάλογος με την ΙΚΑΟ για να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές ούτως ώστε να δούμε τι θα γίνει, ε, ποιες χειραποσκευέ μπορούμε να μεταφέρουμε ε, και να συμπεριλάβουμε εδώ και τις αγορές στο αεροδρόμιο. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μία πιο ε, δίκαιη, πολυτιμή, συγγνώμη, δίκαιη πολιτική τιμών, ούτως ώστε να προσφέρουμε και ποιοτικέ υπηρεσίες. Δεν αρκεί να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση των επιβατών. Αυτό μας είπατε εσείς ε, κύριε Επίτροπε. Δεν με ικανοποιεί αυτή η απάντηση. Σας ε, καλώ να προχωρήσετε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και να κάνετε κάτι παραπάνω από την πληροφόρηση. Ευχαριστώ κύριο Δανέλης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καθώς το τοπίο στις αερομεταφορές της Ευρώπης συνεχίζει να μεταλλάσσεται υπό το βάρος της τιμής του καυσίμου και των μοντέλων χαμηλού κόστους, είναι καταρχήν ευθύνη της ένωσης να διαφυλάξει τα δικαιώματα των επιβατών και ένα δίκαιο πλαίσιο ανταγωνισμού. η εξάπλωση του κανόνα μιας χειραποσκευής παρακάμπτει το πλέγμα των ενισχύ διατάξεων για τα δικαιώματα των επιβατών τα αεροπορικά τέλη και τις κρατικές ενισχύσεις και συνιστά ένα πρόβλημα που οφείλει να αντιμετωπιστεί αφού μεταξύ άλλων πρώτο έχουν προκαλέσει ένα καθεστώς γενικευμένης σύγχυσης στο επιβατικό κοινό οι εκπρόσωποι των καταναλωτικών ενώσεων μιλούν για ένα μείζον πρόβλημα δεύτερο πολλά αεροδρόμια βασίζονται στι πωλήσει των καταστημάτων για σημαντικό μέρο των εσόδων του, γι' αυτά η μονομερής εφαρμογή του κανόνα μια χειραποσκευή πρόκειται για επιζήμια ανατροπή του επιχειρηματικού του μοντέλου και βέβαια για πολλού λόγου επιβάλλεται μια άμεση και εναρμονισμένη εφαρμογή κανόνων και όχι απλά και μόνο μια ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τάιλορ, για ένα λεπτό. Uh, uh. Ευχαριστώ. Είναι πολύ έγκαιρη και εύστοχη η ερώτηση του Πρόεδρου της uh, Επιτροπής Μεταφορών και αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση και με τη ματέωση. Είχαμε τρεις διαφορετικές εκθέσεις που κατέληξαν ε, το 2012 στο, το πρόβλημα που υπάρχει με τις χειραποσκευές και μάλιστα ήμουν ο συντάκτης της πρώτης έκθεσης που αφορούσε την ε, εφαρμογή και λειτουργία των ε, δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών εταιριών και μάλιστα είχαμε σημαντική πλειοψηφία υπέρ τη έκθεση. Ό,τι αφορούσε τι χειραποσκευέ, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα, να προτείνει μέτρα για να εναρμονιστούν οι εμπορικέ πρακτικέ των αεροπορικών εταιριών και να προστατευτούν οι επιβάτε έναντι υπερβολικών περιορισμών και να μπορούν να επιβιβάζουν ένα λογικό αριθμό χειραποσκευών. Εκφράσαμε λοιπόν τι επιθυμίε μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν κατάλαβα καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αφήσει το θέμα στη διακριτική ευχαίρεια των αγορών και σε τελική ανάλυση και των δικαστήριων. Δεν θεωρώ ότι είναι επαρκέ κάτι τέτοιο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση μετά από τι τρει επανειλημμένε εκθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κόσα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιοι ομιλητέ που ζήτησαν το λόγο, δέκα συγκεκριμένα, στα πλαίσια τη διαδικασία Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο σε όλου, αλλά θα πρέπει όλοι να σεβαστείτε το ένα λεπτό. Ξεκινούμε με τον κύριο Μπάνκι. Κύριε Πρόεδρε, ο κανόνας της ενιαίας χειραποσκευής περιορίζει τα δικαιώματα των επιβατών. Δεν έχουμε ενιαίους κανόνες, δεν έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, όταν αγοράζουμε στο ίντερνετ ένα εισιτήριο, δεν ξέρουμε ποιε είναι οι συνθήκε για τι χειραποσκευέ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τι συνθήκε από εταιρεία σε εταιρεία. Συχνά ο επιβάτη τιμωρείται γιατί πληρώνει υπερβολικέ τιμέ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουμε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να επιβάλλουμε ενιαίου κανόνε. Νομίζω ότι αυτό θα είναι προ όφελο και τη λειτουργία των αεροδρομίων, ειδικά των πιο μικρών. Στις 23 Οκτωβρίου του 2012 εγκρίναμε μία γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για αυτό το θέμα και εκεί ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρυθμίσει αυτό το θέμα των χειραποσκευών. Ελπίζω να δοθεί συνέχεια στο αίτημά μας αυτό. Ματούλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε οι Ευρωπαίοι πολίτες, κύριε Επίτροπε, που ταξιδεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ένωση, έχουν ε, διαπιστώσει ότι ορισμένες εταιρείες επιβάλλουν άδικη ε, μεταχείριση ε, για τις χειραποσκευές ε, και εδώ ε, αφορά αυτό και τον αριθμό τους και τις διαστάσεις τους. Ξέρω ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας και θέματα χώρου για τον κάθε επιβάτη και τις αποσκευές του στο αεροσκάφος, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αποτρέψουμε τις εταιρείες να επιβάλλουν καταχρηστικές ρυθμίσεις και απαράδεκτα τέλη και πρόστιμα. Θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες λοιπόν και να γνωρίζουν οι επιβάτες ε, τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν εταιρείε που επιτρέπουν μόνο 7 ε, κιλά να ζυγίζει η χειραποσκευή. Αυτά είναι άδικα. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να σεβόμαστε τα δικαιώματα των επιβατών. Ο κύριος Λάιχτφριτ, ευχαριστώ. Grazie, signora Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, να σας δώσω δύο παραδείγματα. Προσωπικά τα έζησα πριν από λίγο καιρό. Είχα τη ε, χαρά, δεν θα πω το όνομα της εταιρεία, να πετάξω ε, ε, με ένα αεροπλάνο που λέγονταν Πόλη του Βίτεμπεργκ. Ήταν μια πτήση με ανταπόκριση που άργησε πάρα πολύ και με τους επιβάτες, χάος τεράστιο με τις χειραποσκευές. Τελικά καταφέρανε να βάλουν και τους επιβάτες και τις αποσκευές. Λίγο αργότερα πήρα μια άλλη εταιρεία, αντίστοιχα φαινόμενα. Δεν τους επέτρεψαν να έχουν πάνω από μια χειραποσκευή ούτε να μπουκάλι από το duty free. Σκέτο χάος και αυτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες. Τώρα δεν ξέρω, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, να τα γνωρίζουν οι επιβάτες πριν αγοράσουν ε, το εισιτήριο. Εξάρτητα από το αεροδρόμιο, την εταιρεία, θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες σε όλη την Ευρώπη. Και εσείς πρέπει να το φροντίσετε, είναι δικιά σας δουλειά αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι εφαρμόζονται όλο και πιο περιοριστικά μέτρα από τις αεροπορικές εταιρείες, κάτι που δυσκολεύει τη ζωή των επιβατών. Και μάλιστα αυτό οφείλεται όχι μόνο στους κανόνες για τις χειραποσκευές, αλλά και στο θέμα των διαστάσεων των χειραποσκευών και του βάρους των χειραποσκευών. Ο επιβάτης δυστυχώς μαθαίνει για τις διατάξεις αυτές μόνο μετά την επιβίβασή του, όταν είναι ε, αργά δηλαδή, και όταν το μόνο που το απομένει είναι να καταβάλει την επιπλέον χρέωση. Πρόκειται για ένα παράδειγμα συγκαλυμμένων τελών, συγκαλυμμένων επιπλέον χρεώσεων και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί στο θέμα της διαφάνειας των τιμών. Να μην δίνουμε την ευκαιρία σε αεροπορικές εταιρείες να επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις. Κύριο Σιριγκόν. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Γνωρίζουμε και το ακούσαμε επανειλημμένο σήμερα ότι κάποιε αεροπορικέ εταιρείε συνεχίζουν να επιβάλλουν καταχρηστικέ ρήτρε ει βάρο των επιβατών υπό το πρόσχημα τη εξασφάλιση ε, χαμηλών αεροπορικών εισιτηρίων. Έχουν όμω συγκεχημένε ε, τιμέ ουσιαστικά που παραπλανούν τον επιβάτη. Έχουμε περιστάσει όπου μία χειραποσκευή ε, εφαρμόζεται με προβληματικό τρόπο και προκαλεί τις διαμαρτυρίες και τα παράπονα των επιβατών. Μερικές φορές αυτά τα εμπόδια είναι ανυπέρβλητα. Χρειαζόμαστε θέσπιση νομοθεσίας με σαφή και διαφανή ενημέρωση. Επίγει η λήψη μέτρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να εξασφαλιστεί η σωστή πληροφόρηση και η διαφάνεια για τον υπολογισμό της τιμής του αεροπορικού εισιτηρίου εισιτηρίου. Επίσης, ε, τα μέτρα για τη χειραποσκευή θα πρέπει να διευκρινιστούν, να ξέρει ο επιβάτης τι δικαιούται να μεταφέρει στο αεροπλάνο. Θέλουμε εξασφάλιση των δικαιωμάτων, ασφάλεια, κατάργηση των καταχρήσεων και φυσικά κάποιες εγγυήσεις και για τους επιβάτες και τις αεροπορικές εταιρείες. Ο κύριος Κλίντς. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι κόπτεται για την προστασία των καταναλωτών, ε, τον δίκαιο ανταγωνισμό και τη διαφάνεια. Στην πράξη τελείω διαφορετικά τα θέματα ε, για αυτά που μας απασχολούν. Έχουμε ο στην την εμπειρία του από αεροπορικέ εταιρείε. Μεγάλες διαφορές έχουν ε, και μάλιστα στον ορισμό του τι εστί αποσκευή και τι χειραποσκευή και τι μπορεί κανεί να πάρει μαζί του. Και οι χαμηλού κόστου εταιρείε τεράστια αυθαιρεσία. Ξέρουμε μια κυρία από τη Λιόν που την ανάγκασαν να βγει από το αεροπλάνο μόνο γιατί αρνήθηκε ε, να ε, δώσει είτε την τσάντα τη είτε ένα ποτό που είχε αγοράσει σε ένα κατάστημα του αεροδρομίου. Δεν γίνεται αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών το τελευταίο διάστημα. Μα θεωρούν γραφειοκράτε και ε, εχθρικού προ τον καταναλωτή. Κάντε κάτι επιτέλου, αξιοποιήστε την ευκαιρία και δώστε τα δικαιώματα στου πολίτε που έχουν. Ο κύριος Μπάνιον. Ο κύριος Μπάνιον. Εγώ καλωρίζω, καλωσορίζω αυτή την προφορική ερώτηση. Είναι περίπλοκη η κατάσταση τώρα στις πύλες εισόδου. Ε, το πρόβλημα είναι ότι δεν ε, ενημερώνται σωστά οι επιβάτες. Συχνά υπάρχουν καυγάδες μεταξύ επιβατών και προσωπικού. Χρειαζόμαστε μια κάποια συνέπεια. Επίσης, ε, Υπάρχει πρόβλημα με τι ε, δραστηριότητε λιανεμπορίου στα αεροδρόμια. Το πρόβλημα εδώ είναι οι περιορισμοί που επιβάλλονται. Συμφωνώ με την Κομισιόν ότι κάποια διαφοροποίηση ε, προωθεί τον ανταγωνισμό. Να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά όχι πολύ αυστηροί όμω. Θέλουμε ένα ελάχιστο ανώτατο όριο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ενιαίο όριο, γιατί σίγουρα είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες των εταιριών low cost από τις υπόλοιπε κανονικές εταιρείε. Επίσης είναι διαφορετικές οι ανάγκες των εταιριών οι οποίες πετάνε σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ε, επομένως θα πρέπει να παρέμβουμε λίγο και με λογικό τρόπο. Μέσνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στην Ευρώπη έχουμε ρύθμιση για ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών. Αυτό είναι και έμβλημά μας. Ε, και δεν θέλουμε υπερβολικές ρυθμίσεις, αλλά ένα λογικό πλαίσιο. Αυτό που έχουμε σήμερα κατά την άποψή μου αδιαφανές, ε, ε, αυθαίρετο και εχθρικό προς καταναλωτές. Να σας πω ότι έζησα εγώ, έχω πολλά παραδείγματα με μια εταιρεία χαμηλού κόστους ταξίδευα στην Ευρώπη. Είχα μια μικρή τσάντα μαζί μου και την τσάντα μου. Και σχεδόν δεν με άφησαν να επιβιβαστώ. Είχαν ένα στάντ για να δώσει τις αποσκευές, ε, τις έριχνες εκεί μέσα. Τους έδειξα ότι έχω μια μικρή αποσκευή και μια μικρή χειραποσκευή και μου είπαν θα πληρώσεις ή θα φύγεις. Μεγάλο ψυχόδραμα το ήξερα, αλλά το δοκίμασα για να δω τι θα συμβεί. Υπάρχουν άλλοι επιβάτε που δεν το γνωρίζουν καν και δεν ξέρουν και τα δικαιώματά τους. Δεν επιτρέπονται αυτέ οι καταστάσει. Εγώ είμαι πάντα κατά της υπερβολικής ρυθμίση, αλλά εδώ χρειαζόμαστε λογικού κανόνες. Η κυρία Κάντεμπαχ. Η κυρία Κάντεμπαχ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έχουμε ζήσει πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι είναι απαραίτητη μια λογική ρύθμιση, ε, αλλά να ανταποκρίνεται και στην πράξη, γιατί δεν έχει νόημα να φτιάξουμε κανόνες που τελικά ε, παρακάπτονται από παραθυράκια, επιτρέπουν επιπλέον κόστο και μεγαλύτερη αδιαφάνεια στην ε, τιμολόγηση του εισιτήριου. Θα σα παρακαλούσα να συζητήσετε με ανθρώπους που δεν είναι μόνο business επιχειρηματίε αλλά είναι η πρώτη, πρώην τρίτη θέση, αν θυμάστε, που υπήρχε παλιά, που έχουν παιδιά, που έχουν ε, αποσκευέ και δεν είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στο αεροπλάνο και προσπαθούν να μπουν με τις αποσκευέ τους και δεν υπάρχει χώρος πουθενά να βάλουν τα πράγματά τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν λογικούς κανόνες. Και ποιοι είναι οι λογικοί δεν μπορώ να βάζω στα παιδιά μου πέντε πουλόβερ και πέντε ζακέτες γιατί ζακέτε ζεστή σε μία χώρα κρύα και δεν έχω χώρο στις αποσκευές μου. Ε, καθημερινά τα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Αλλά αυτό να μην οδηγήσει σε μια χωρα κρυα και δεν εχω χωρο στι αποσκευε μου ε καθημερινα τα βλεπουμε αύξηση τη τιμή του εισιτηρίου. Κυρία Μπιλμπάου, ευχαριστώ. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη συμφωνία σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς που πλήττουν σαφώς τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιρεών που αναγνωρίζονται από την κοινοτική νομοθεσία και προκαλούνται ζημιές και στα καταστήματα των αεροδρομίων. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις αυθαιρεσίες. Όσο περιμένουμε όμως μεταρρυθμίσεις ή εναρμόνιση που επανειλημμένως ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια διαδικασία που θα είναι αρκετά χρονοβόρα, στο μεταξύ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, να ενισχύσουμε τα μέτρα ελέγχου, να ασκήσουμε πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες και να αυξήσουμε τις κυρώσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση που εφαρμόζουν τέτοιες παραπλανητικές ή απατηλές πρακτικές. Πρακτικές. Ερωτώ λοιπόν τον Επίτροπο. Θεωρείτε ότι είναι εύστοχη μια ιδέα διοργάνωσης ε, ενημερωτικής εκστρατείας για να ενημερωθούν οι επιβάτες για τις πρακτικές αυτές. Επίσης, ε, ίσως ε, με ψηφιακό τρόπο θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε τα αεροδρόμια για το τι δικαιώματα ελέγχου έχουν απέναντι σε αυτές τις αεροπορικές εταιρείες. Γιατί και οι επιβάτες και τα αεροδρόμια πλήττονται μερικές φορές από καταχρηστικές πρακτικές. Μπορείτε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είστε ε, έτοιμοι, πρόθυμοι να οργανώσετε τέτοια ενημερωτική εκστρατεία. κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, την τελευταία δεκαετία η μετακινήσεις επιβατών μέσω των περιφερειακών αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 84% και το 90% των δικτύων αεροδρομίων είναι ουσιαστικά περιφερειακά αεροδρόμια. Επαναλαμβάνω, τελευταία δεκαετία έχουν ενισχυθεί αισθητά οι μεταφορές μέσω τέτοιων αεροδρομίων. Πρέπει επιτέλους ε, να παταχθούν ε, οι καταχρηστικές πρακτικές των αεροπορικών εταιριών. Χρειαζόμαστε κάποια μέτρα για εναρμόνιση εμπορικών πρακτικών των αεροπορικών εταιριών. Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε τους επιβάτες ε, κατά καταχρηστικών πρακτικών και περιορισμών. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στους πολίτες να μπορούν να, μεταφέρουν ένα λογικό αριθμό χειραποσκευών στο αεροπλάνο. Δραστικοί περιορισμοί τη μια χειραποσκευή που εφαρμόζουν κάποιε αεροπορικέ εταιρείε ε, αποτελεί κατάφορη παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Επίση, τα τέλη που επιβάλλονται μερικέ φορέ είναι υπέρογκα, δυσανάλογα υψηλά και διαταράσσουν και την πολιτική διαφάνεια που πρέπει να ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον καθορισμό των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων. Τελείωσε εδώ το Catch the Eye. Ο Επίτροπο Δεχούχτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, Ευρωβουλευτές για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο αριθμός των παρεμβάσεων δείχνει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το θέμα και θα συνεχίσω να δουλεύω επί πολιτικών που υποστηρίζουν τα συμφέροντα των επιβατών καθώς και μηχανισμούς, ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στην νομοθεσία. Όπως είπα στις εγωικές μου παρατηρήσεις, πολύ σύντομα θα αναθεωρήσουμε τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών στη σχετική νομοθεσία θα παρουσιαστεί από τον Επίτροπο κύριο Κάλλα αυτό το νέο νομοθέτημα το πρώτο εξάμεινο του 2013 και τότε θα είναι νομίζω και η κατάλληλη ευκαιρία για να συζητήσουμε πιο ενδελεχώ όλα αυτά τα σημεία τα οποία σχολιάστηκαν σήμερα τους Ευρωβουλευτέ. Τούτου λεχθέντος νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό. Θέλετε περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, γιατί μερικές φορές ε, οι επιβάτες αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Θέλω να προσθέσω ότι ο επίτροπο Κάλλας ήθελε και ο ίδιος να συμμετάσχει σήμερα προσωπικά στην συζήτηση, αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξε η ημερήσια διάταξη αυτής της εβδομάδας και τον εμπόδισε να παραστεί προσωπικό. Πάντως θα του διαβιβάσω όλα τα σχόλια τα οποία κάνατε και όταν συζητήσουμε το νομοθέτημα για τα δικαιώματα των επιβατών στι αεροπορικέ εταιρείε θα μπορέσει και ο ίδιο να τοποθετηθεί προσωπικά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τελείωσε αυτή η συζήτηση. Τώρα με βάση την ημερήσια διάταξη περνάμε στην προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τον καονισμό σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της καταγωγής ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες.